Πρώτη ψηφοφορία επί ε, τη αιτήσια εκθέσεω του Δημοσιολαβητή για το 2010. Ε, μία ψήφο υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται η εκθέση Ιώτοβα. Συγχαίρω την εισηγήτρια. Επόμενο θέμα. Έκθεση Αντζελίλη. Σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία. Πρόταση οδηγία. Τροπολογία παριθμών 1 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψήφι υπέρ της πρότασης Κομισιόν. Κατά αποχές εγκρίνεται η πρόταση Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Πολλά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Επόμενο θέμα. Ψηφοφορία τη ω Λάμπερτ για τι ελάχιστε απαιτήσει για την αναγνώριση και το καθεστώ των υπηκών τρίτων χωρών ή των ανηθαγενών ω δικαιούχων διεθνού προστασία. Πρώτο πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η πρόταση λοιπόν της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Και τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, τροπολογία 2, χωρίς ψηφοφορία, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος συνολικά με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγητριά μας. Επόμενο θέμα είναι η πρόταση ψηφίσματος εκ μέρους της ομάδας ε, της ΓΚΟΕ για γνωμοδότηση του δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα της συμφωνίας PNR μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστραλίας. Ψηφίζουμε την πρόταση αυτή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ξεκάθαρα και περνάμε στο επόμενο θέμα. Έκθεση Intveld. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστραλίας για, την, για τα στοιχεία επιβατών PNR. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ονομαστικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και συγχαίρουμε την συγκήτρια. Επόμενο θέμα. Ψηφοφορία επί 7 προτάσεων ψηφίσματος για την κατάσταση στην Αίγυπτο και στη Συρία, ιδίως όσον αφορά τις χριστιανικές κοινότητες. κύριος Μάουρο νομίζω έχει μια προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας διαβάσω σύντομα μια τροπολογία τεχνική φύση που ήδη έχουμε συμφωνήσει με τις άλλε ε, ομάδες. Είναι στο σημείο 5. Καλεί τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να συμμορφωθούν αυστηρά προς την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων. Ε, καλεί τον Αντιπρόεδρο της, της, την, της Επιτροπής, την είπα το εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την ε, Πολιτική Ασφάλεια, την Κάθριν Άστον, ώστε να ζητήσει από τα κρατημέλη να εφαρμόσουν και να συμμορφωθούν προς απαιτήσεις τη κοινής θέσης. Αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κοινή πρόταση ψηφίσματος συνολικά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία. Έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία. Παράγραφο 2. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα ήθελα να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 2. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Παράγραφο 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Χωριστή ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. λογική σκέψη. Σι γάμα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κοινή πρόταση ψηφίσματος συνολικά ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στην πρόταση ψηφίσματος Επιτροπής Περιβάλλοντος για την απειλή της ε, μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι το, στην παράγραφο 32 θα επανεισαχθεί το αρχικό κείμενο όπως ψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή. επιτροπή. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 7. Παράγραφος 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Προτιμώ να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Επίσης μονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της πρότασης περ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 Ερχόμαστε τώρα στις επεξεγγίσεις ψήφου. Πρώτα ο κύριος Σιλβέστρης. Για την έκθεση ε, Ιωτόβα.